Εδώ τελειώνει το πρώτο τμήμα της συνεδριάσής μας και τώρα το επόμενο θέμα κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Μεταφορών για, του, της οποίας τον πρόεδρο ευχαριστώ για την υπομονή του Σας καλωσορίζω καθώς και τους συναδέλφους και τους καλεσμένους και τους ομιλητές και τις ομιλήτριες που είχαν την ευγενή καλοσύνη να προσέλθουν σήμερα στη συνεδρίασή μας. Το θέμα είναι το Connecting Europe και θα υπάρξει συμπροεδρία των δύο επιτροπών. Η κοινή αυτή συνεδρίαση περιλαμβάνει και δημόσια ακρόαση για το Connecting Europe. Το θέμα είναι πώς θα κινητοποιήσουμε καλύτερα τους χρηματικούς μας πόρους για να συμπληρωθεί αυτό το φιλόδοξο διεθνές πρόγραμμα υποδομών. Θα τεθούν και πρακτικά προβλήματα θα συζητηθούν. Θα προεδρεύσω στην αρχή εγώ και μετά ο Μπράιαν Σίμψον. Έχουμε εδώ σήμερα μερικούς εξαιρετικούς ομιλητάς και θα τεθούν και ερωτήματα από τους συναδέλφους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι αυστηρότατοι με το χρόνο ομιλίας μας. Παρακαλώ τους παρουσιαστές να περιοριστούν σε 10 λεπτά και οι ερωταπαντήσεις θα έχουν πολύ λίγο χρόνο γιατί στο σύνολο έχουμε μόνο 20 λεπτά για τις ερωταπαντήσεις. Ένα λεπτό κάθε βουλευτής. Άρα να είναι πολύ στοχευμένες οι ερωτήσεις παρακαλώ. Πρώτος ομιλητής, Μαρκ Μπράιερ. Και θα μας μιλήσει για τις ελλείψεις που έχει διαπιστώσει. Καλημέρα σας. Ήρθα σήμερα να σας μιλήσω για τις κυριότερες χρηματοδοτήσεις really ναι. για τις υποδομές. Η αγορά αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην Ευρώπη και όταν σημειώθηκε η πρώτη κρίση σχεδόν καταστράφηκε η αγορά αυτή. Αυτή τη στιγμή λόγω των απαιτήσεων της Βασιλείας 3 υποχωρεί κάπως το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί θεσμικοί επενδυτές αλλά δεν χρησιμοποιούν και τόσο πολύ τις λεγόμενες brownfield infrastructures. Need to be addressed, and they are very specific. Uh, what I'm going to tell you today. Σήμερα δεν θα σας πω τίποτα δύσκολο. Αν και θα εισέλθω σε λεπτομέρειες. And what are the problems of borrowers and what are the problems of investors? Τα ομόλογα έργου είναι κάτι απαραίτητο Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι οι δανειστές δεν έχουν μεγάλο βάθος και αυτό είναι για αυτούς πρόβλημα. Τα έργα χρειάζονται επενδύσεις. Μερικές τράπεζες δεν χορηγούν εύκολα δάνεια και γι' αυτό μειώνεται γενικά η χρηματοδότηση. Ακριβένει η επένδυση και αυξάνεται ο κίνδυνος. Πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες φούσκες. Η λύση του προβλήματος αυτού των δανειστών των δανειζομένων μάλλον, των δανειοληπτών, είναι να υπάρχει σταθερό επιτόκιο μακροπρόθεσμο και να, μειωθούν, να μειωθεί το κόστος. Η απλοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας πρέπει να γίνει, αλλιώς οι δανειολήπτε δεν θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το πρόβλημα των επενδυτών είναι καλά γνωστό στις αγορές, ίσως όχι εδώ, αλλά από τους γνώστες σαν και εμένα είναι κάτι πολύ κοινό. Δεν έχουν και μεγάλη όρεξη για σημαντικές επενδύσεις γιατί δεν υπάρχει ομογενοποίηση των επιτοκίων φάνηκε αυτό και από την πρόσφατη κρίση και ανησυχούν για τις μεμονωμένες επενδύσεις one-off που δεν ανταποκρίνονται όμως και ακριβώς στα συμφέροντά τους. Η λύση του προβλήματος αυτού είναι απλούστατη κατεμένα. Πρέπει να υπάρχει σωστή επιτήρηση και δόμηση ώστε να οι επενδυτές να θέλουν να αγοράσουν τέτοιου είδους ομόλογα να έχουν την εμπιστοσύνη ότι ακόμη και με σε δύσκολες συνθήκες θα εφαρμοστούν τα συμπεφωνημένα με ομοιόμορφο τρόπο να υπάρχει κάποια τυποποίηση στην πληροφόρηση ώστε να μπορούν οι επενδυτές κάθε τρίμηνο να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την πρόοδο των επενδύσεών τους και να μπορούν και να αντιδράσουν όταν κάτι πάει στραβά. Εδώ βλέπετε κάτι που μοιάζει σαν πολύπλοκο αλλά που αφορά κάτι πολύ απλό στην αγορά σήμερα. Δηλαδή τα προβλήματα και τις λύσεις που μόλις συζήτησα μέσα στην ίδια δομή. Δηλαδή η δομή αυτή είναι εκείνη που σχεδιάσαμε πριν από τρία χρόνια και για την οποία συνεργαστήκαμε και με την ΕΤΕ. Τώρα, ποιες δοσοληψίες υπάρχουν, είναι διαθέσιμες. Υπάρχουν αυτές που είναι χαμηλού κινδύνου και υψηλού κινδύνου. Οι επενδυτές που αγοράζουν ομόλογα πρέπει και τους δύο αυτούς τομείς να τους βλέπουν ρητά να βλέπουν ρητά τα ωφέλη αλλιώς δεν θα αγοράσουν τα ομόλογα βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν πολλές δοσοληψίες στον χαμηλού κινδύνου τομέα Υπάρχουν και μερικές που είναι μεταξύ των δύο. Ο τρόπος αποτίμησης των δύο τύπων κινδύνου αφορά την δόμηση των ομολόγων των ίδιων. Υπάρχουν μερικά προβλήματα σε αυτού του είδους τα ομόλογα που προσπαθούμε όλοι να τα λύσουμε για μεγαλύτερων διαστάσεων προγράμματα δουλεύουν καλύτερα τέτοια ομόλογα. Είναι μεγάλος κίνδυνος για τους επενδυτές ορισμένων ε, τύποι ομολόγων. Τα κρατικά χρέη είναι άλλος τομέας. ως προς τη δυνατότητα πώληση ομολόγων του χρέους και από τα κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρωζώνη είναι οι κανόνες για τις πραμήθειες που φαίνεται ότι δεν δουλεύουν όπως θα έπρεπε. Τέλος, θέματα... Uh, insurance companies and θέματα λειτουργίας των ε, συνταξιοδοτικών ταμείων ας πούμε είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Φαίνεται λοιπόν ότι τα υψηλότερου κινδύνου προγράμματα έχουν και υψηλότερη τιμή και κόστος. Συμπεράσματα. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα δανειοδότησης στην Ένωση, κυρίως ε, για τις ασφαλιστικές εταιρείες και για τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι η δανειοληψία σημαίνει ότι οι επενδυτές θέλουν να αγοράζουν ομόλογα αλλά όχι κανονικά δάνεια. Καλά δομημένα δάνεια τώρα είναι κάτι το τελείως βασικό για να λυθούν τα προβλήματα της Ένωσης στο μέλλον. Αυτά τα ομόλογα έργο πρέπει να έχουν εγγυήσεις, αυξημένες εγγυήσεις για να υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθούν γρήγορα. Και μόνο τότε θα μπορέσει να επιταχυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα για τα ομόλογα έργου είναι ένας καλός καταλήτης για όλα αυτά. Πρέπει η αγορά αυτή να προωθηθεί, αλλά οι ιδιωτικέ δανειοδοτήσεις ή δανειοληψίες θα χρειαστούν και αυτές μαζί με τα ομόλογα έργου. λόγω των μαζικών αναγκών χρηματοδότηση που έχει η Ευρώπη για τις υποδομές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την τοποθέτηση αλλά και για τον σεβασμό του χρόνου. Ο κύριος Ντέιβιτ <coughs> Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα για την χρηματοδότηση των υποδομών στο τομέα της ενέργειας και τον ρόλο που οι ρυθμιστικές αρχές διαδραματίζουν όσον αφορά τις υποδομές και την χρηματοδότηση. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτός και πρέπει να εξετάζεται μέσα στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων για την Connecting Europe Facility, το μέσο της διασύνδεσης ε, της Ευρώπης και την χρηματοδότηση όσον αφορά τη νομοθετική πρόταση που πρέπει να ε, πούμε ότι βρίσκεται υπό εξέταση τώρα εδώ. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι κανονικά και ιστορικά οι υποδομές στον ενεργειακό τομέα καλύπτονται μέσω των ε, τιμολογίων των δικτύων. Εκείνοι που το χρησιμοποιούν πληρώνουν τα τιμολόγια αυτά και φυσικά και οι πάροχοι υπηρεσιών καλύπτουν έτσι τις δαπάνες τους ε, με την ίσπραξη αυτών των εσόδων. Τι σημαίνει αυτό σε σχέση με την υποδομή. Η ασφάλεια που έχουν ε, οι εταιρείες που απορρέει από τις συμβάσεις και τα συμβόλαια από τους καταναλωτές που πληρώνουν αυτά τα τιμολόγια δίνουν μεγάλη πιθανότητα να καλύπτονται αυτά τα έξοδα και υπάρχει χαμηλός κίνδυνος πιθανότατα. Αυτή η διαδικασία λειτουργήσε πολύ καλά στο παρελθόν και χρηματοδότησε πολλές υπόδομες. Όμως δυστυχώς σήμερα βλέπουμε νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και φυσικά έχουμε και την χρηματοοικονομική κρίση και τις ε, κλιματικές αλλαγές, ε, νέες προκλήσεις, νέες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια στον ε, ενεργειακό τομέα και την ασφάλεια εφοδιασμού. Όλα αυτά απαιτούν νέα μέτρα υποδομών στην Ευρώπη για να έχουμε ένα ασφαλές πλαίσιο και χαμηλών εκπομπών ρήπων στην αγορά ενέργειας. Τώρα, τούτων λεχθέντων, τα θεμέλια της χρηματοδότησης για το μέλλον και η συντριπτική πλειοψηφία της χρηματοδότησης που απαιτείται για τις υποδομές στον ενεργειακό τομέα θα προέλθει από αυτή την ρύθμιση όσον αφορά τα έσοδα από τιμολόγια και τις τιμές. Φυσικά θέλουμε να διευκολύνουμε οι επενδυτές να έχουν πρόσβαση στις πιο αποτελεσματικές μορφές κεφαλαίων και ως ρυθμιστές, ρυθμιστικές αρχές είναι ευπρόσδεκτες οι προτάσεις να έχουμε καινοτόμες προτάσεις για τους επενδυτές που θα είναι οι καινοτόμες προτάσεις στη διάθεσή τους. Αν δει κανεί το συνολικό πλαίσιο όσον αφορά την άμεση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια 9,1 δις ευρώ φαίνεται ότι είναι μεγάλο ποσό όμως μέσα στο πλαίσιο των τεράστιων κονδυλίων που χρειάζονται για το, για το μέλλον στην Ευρώπη για τις υποδομές είναι σχετικά μικρό ποσό. Δεν θα είχα αντίρρηση να το έχω αυτό το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό μου βέβαια εγώ, αλλά στο πλαίσιο των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης είναι χαμηλό, μικρό ποσό αυτό. Επόμενο τώρα. Φυσικά όταν οι επενδύσεις θα έχουν γίνει στις υποδομές πρέπει να μεριμνήσουμε και να δούμε ποιος θα πληρώσει για όλα αυτά. Και υπό το πνεύμα των ρυθμιστών θεωρούμε ότι εκείνοι οι οποίοι υποφελούνται από τις υποδομές θα πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι θα πληρώσουν το αντίτιμο. Λοιπόν, αν οι καταναλωτέ σε μια χώρα εποφελούνται από χαμηλότερε τιμέ σαν αποτέλεσμα επενδύσεων στι υποδομέ, εκείνοι λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να πληρώσουν για το κόστο αυτών των υποδομών. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα εκείνη θα πληρώσει όπου θα δημιουργηθούν υποδομέ υποχρεωτικά. Πρέπει να έχουμε μηχανισμού λοιπόν που θα λειτουργήσουν ώστε το κόστο των υποδομών να επιμερίζεται δίκαια σε εκείνου που θα συμμερίζονται και θα συμμετέχουν σε αυτό το κόστος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποια ωφέλη σε σχέση με το σύνολο των καταναλωτών. Μείωση στις εκπομπές ρήπων π.χ. Αν έχουμε επενδύσεις ε, σε σχέση με αυτόν τον τομέα όλοι οι κατανάλωτε στην Ευρώπη θα υποφεληθούν. Όχι μόνο εκείνοι στη χώρα των οποίων οι υποδομέ αυτέ θα διασφαλιστούν και πρέπει οι μηχανισμοί για το αντίτιμο το οποίο θα εισπράτεται να είναι δίκαιοι. Και εδώ έχουμε τον ρόλο των ρυθμιστικών αρχών λοιπόν και χαιρόμαστε για το ότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επομιστεί αυτόν τον ρόλο συγκεκριμένα. Τούτων λεχθέντων όμως τώρα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου κάποια καλά εγχειρήματα και πρωτοβουλίες με σαφή ωφέλη μπορεί να μην στεφθούν με επιτυχία. Ίσως κιόλα επειδή οι κίνδυνοι είναι υπερβολικά υψηλοί και ίσως επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί αρκετοί όσον αφορά τους εποφελούμενους που να επαρκούν για να καλυφθούν τα κόστη. Το βλέπουμε αυτό και στην Ανατολική Ευρώπη, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου οι αγορές δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένες όπως σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Και αυτό φυσικά οδηγεί στην διαχείριση των κινδύνων, αντιμετώπιση των κινδύνων, των επενδυτικών κινδύνων. Τώρα τούτο ακριβώς είναι, αυτό αφορά τον καθορισμό του πώς θα καθορίζουμε, ποια εγχειρήματα είναι εκείνα, ποιες πρωτοβουλίες είναι εκείνες που θα ε, τύχουν προτεραιότητας από τι τις πολλές προτάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία μπορεί να καλύπτεται με τα τιμολόγια, αλλά το να βρούμε εκείνες τις πρωτοβουλίες που αξίζουν, την υποστήριξη, αξίζουν υποστήριξης και ενίσχυσης για να στεφθούν με επιτυχία το να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ποιε από αυτές τις πρωτοβουλίες θα τύχουν προτεραιότητας και θα υποστηριχθούν θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα προγράμματα να μην την χάνουν κάποιας καθυστέρησης όταν θα έχουμε το θέμα της αξιολόγησης και απόφασης ποια προγράμματα θα πρέπει να ενισχυθούν. Ένας τρόπος για να παράσχουμε υποστήριξη είναι οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν πολλαπλά. Πολυσχηδός. Μία προσέγγιση είναι να δοθεί ευκαιρία στους καταναλωτές σε κάποιες περιπτώσεις να ανακουφίσουν τους κινδύνους των επενδυτών. Ένας μηχανισμός, μια δυνατότητα που υφίσταται είναι οι εξαιρέσεις των ε, τρίτων για τρίτους εμπλεκόμενους και ένα στοιχείο ε, κινδύνου έτσι μπορεί να μετακυλίεται στους ε, καταναλωτές. Ένα άλλο ε, μέσο είναι κίνητρα για τις ε, ρυθμιστικές ε, αυτές πρωτοβουλίες όπου θα υπάρχει επιστροφή, μέρισμα αυξημένο με σταθερά καθορισμένους στόχους στη στοχοθέτηση. Παράδειγμα, επιτάχυνση κάποιου είδους επενδύσεων. Επιτάχυνση αν είναι αποφασιστικής σημασίας και στέφεται με επιτυχία, τότε θα έχουν αυξημένο μέρισμα ως επιστροφή. Αλλά αν δεν πετύχουν τους στόχους και είναι, ε, ε, έχει ένα μεγαλύτερο ε, ρυθμό βραδύτητας, τότε θα είναι ισχνότερα τα μερίσματα. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν ώστε ανάλογα με τις ανάγκες να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης δεν υπάρχει μία ρύθμιση που να είναι ικανή και ικανοποιητική για όλες τις πρωτοβουλίες. Εμείς ως ρυθμιστικές αρχές θεωρούμε ότι η διαχείριση των κινδύνων πρέπει να είναι κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες των ατομικών πρωτοβουλειών και εγχειρημάτων. Και ο ρόλος των ρυθμιστών, ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά τρίτα μέρη και τι τις πρωτοβουλίες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Και έχουμε και την ε, ανησυχία ότι κάποιες συγκεκριμένες δεσμευτικές ε, ε, ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι θέμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτροπολογίας, Comitology, όσον αφορά τη, το σχεδιασμό και τις προτάσεις. Τούτων λεχθέντων όμως, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο όπως μπορεί να ισχύσει στο τρίτο πακέτο, μπορεί να εφαρμοστεί και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Αλλά θα υπάρξουν και κάποιοι τομείς όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί να μην είναι επαρκέ ομάδες. Βλέποντας τώρα το πώς θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τα ποια τέτοια σχέδια και προγράμματα θα απαιτούν πρόσθετα μέτρα, θα πρέπει να έχουμε μια ανάλυση, μια αξιολόγηση κόστους-οφέλους, ώστε να βλέπουμε επιμέρους ποσοτικά και καθορίζοντας τα ε, κριτήρια αυτά το τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Να δούμε ποια προγράμματα θα πρέπει, ποια σχέδια θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα και ποια θα είναι επιλέξιμα για υποστήριξη, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν τα, ή να προχωρήσει η πλειοψηφία των προγραμμάτων χωρίς να υπάρχει βραδύτητα ή επιβράδυνση λόγω της ε, διαδικασίας αξιολόγησης. Πιστεύουμε ότι αν τα ωφέλη είναι σαφή, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες για την βιωσιμότητα χρησιμότητα της χρηματοδότησης ενός προγράμματος, ενός σχεδίου, τότε πρέπει να εξετάσουμε αν περαιτέρω μέτρα θα πρέπει να ε, υιοθετηθούν για την βιωσιμότητα. Το κρίσιμο σημείο εδώ είναι η σαφήνεια και στην λήψη απόφασης να δούμε ποια προγράμματα εντάσσονται σε ποια κατηγορία και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συμπεραίνω, οι ρυθμιστικές αρχές για τα θέματα ενέργειας υποστηρίζουν την επιτάχυνση και την ανάγκη να προχωρήσουμε στις ε, επενδύσεις στις υποδομές. Fast track είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε στεναρά. Χρειαζόμαστε σαφή κριτήρια για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ενεργειακών προγραμμάτων και για εκείνα τα προγράμματα που χρειάζονται και πρόσθετη χρηματοδότηση. Πιστεύουμε ότι εκείνα που δεν θα πρέπει να τύχουν υποστηρίζουν είναι εκείνα τα προγράμματα που είναι ήδη βιώσιμα εμπορικά. Και έτσι λοιπόν πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εκείνα τα προγράμματα πρέπει επίσης να εντοπίζονται ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάσης ο οποίος είναι τμήματάρχης στους γαλλικούς σιδηροδρόμους. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω που το δίκτυο υποδομής των σιδηροδρομικών υποδομών προσπάθησε να αναπτύξει σήμερα, μέσα, μέχρι σήμερα μέσα από μεγάλα σχέδια μέσω των οποίων προσπαθήσαμε να Έχουμε ιδιωτική χρηματοδότηση ή προχρηματοδότηση. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το ένα σχήμα και όχι το άλλο. Θα σταθώ σε τέσσερα συμβόλαια μεταξύ, που συνάψαμε μεταξύ 2007-2008 έχουμε τρία ε, ήδη υπογεγραμμένα και ένα τοπίο όπου να είναι θα κλείσει. Μεταξύ αυτών των σχεδίων τα τρία αφορούν ε, τη δημιουργία σίδηροτροχιών υψηλής ταχύτητας, 300 χιλιόμετρα μεταξύ Τουρ Μετά έχουμε ένα άλλο συμβόλαιο που είναι και το πρώτο το οποίο υπογράψαμε, είναι το σχέδιο GSM σιδηρόδρομη και αποτελεί μία συνιστόσα του, του διαλειτουργικού ευρωπαϊκού συστήματος RTMS. Θα έχουμε 15 δισεκατομμύρια εκατομμύρια στο χαρτοφυλάκιο αυτού του σχεδίου με ιδιωτική χρηματοδότηση ή ιδιωτική προχρηματοδότηση όταν θα έχουμε ένα σχήμα συμβολέου συνεργασίας Οι ουσιαστικές διακρίσεις υπάρχουν πολλές. αφορά στην προσέγγιση που έχουμε για τη μεταφορά κινδύνου. Σε μια συμφωνία συνεργασίας, ένα συμβόλαιο συνεργασία, ο δικαιούχο αμείβεται για την παροχή ε, της υποδομής την οποία κατασκευάζει και συντηρεί. Χωρίς τον ε, κίνδυνο της ε, κυκλοφορίας, όταν εμείς υλοποιούμε ένα σχέδιο σαν αυτό τη σύνδεσης Λεμό Ρεν ή σαν αυτό της παρακαμπτηρίου του Μομπελιέ, ο διαχειριστής του δικτύου είναι αυτός που διαχειρίζεται την διακίνηση. Όταν έχουμε παραχώρηση όμως, ο κίνδυνος διακίνησης μεταφέρεται. Πρόκειται για ένα στίχημα. Δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μία σιδηροδρομική παραχώρηση με μεταφορά κινδύνων διακίνησης και το ρίσκο της ε, κυκλοφορίας είναι πολύ μικρότερο από ότι στους αυτοκινητοδρόμους. Για την σύλληψη, ε, κατασκευή και συντήρηση υπάρχει λίγη διαφορά μεταξύ των δύο σχημάτων. Έχουμε σε περίπτωση παραχώρησης ιδιωτική χρηματοδότηση συν ε, επιδοτήσεις για τη συντήρηση. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε ε, παραχώρηση χωρίς ε, επιδοτήσεις για συντήρηση. Είναι πολύ δύσκολο στους αυτοκινητοδρόμους και παραμένει δύσκολο και στους σιδηροδρόμους. Αλλά πέρα από την επενδυτική επιδότηση, η παραχώρηση εξισορροπείται από μόνη της μέσα από την δασμολογική ε, παροχή όταν τίθεται σε λειτουργία. Οι επιδοτήσεις ε, επιστρέφονται κατά την διάρκεια του συμβολέου. Μετά έχουμε υπολογισμό του ρίσκου, για το κατά πόσο δηλαδή ο... αυτός ο οποίος έχει λάβει την εκχώρηση μπορεί να διατηρήσει. Στον ιδιωτικό τομέα βλέπετε λαμβάνουμε υπόψη ε, το ρίσκο σε μεγάλο βαθμό. Με τη διαφορά που βλέπετε στο, στο σχεδιάγραμμα, όπου έχουμε διαφορές ε, μεταξύ συνεργασίας ή εκχώρησης. Τώρα, για τη χρηματοδότηση των δύο σχεδίων, η γραμμή μεταξύ Τουρ και Μπορντό και η γραμμή της Ρένα Βλέπετε ότι έχουμε επιδοτήσεις επενδυτικές και τα υπόλοιπα καλύπτονται από ίδιους πόρους και συγχρηματοδότηση το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από ενδιάμεσες δαπάνες συνολικά στην όλη γραμμή εκχώρησης. Αν στην εκχώρηση αν ο δικαιούχος αμείβεται μέσα από τα διόδια σε περίπτωση συνεργασίας έχουμε προχρηματοδότηση αλλά και νίκια, ή δασμούς, υπάρχει πολλή ορολογία για να περιγράψουμε αυτού του τύπου τα έσοδα. Στα στις δύο μορφές συμβολέου που χρησιμοποιούμε. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση μέσα από την απόδοση και έχουμε και ένα πίλοταζ μέσα από τα συμβόλαια εκχώρησης. Θα τελειώσω με ένα τελευταίο σημείο. Δεν έχουμε ακόμη τεχνολογικά σχέδια για να τα χρηματοδοτήσουμε σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, αλλά για τις γραμμές τρένων υψηλής ταχύτητας εμείς ε, βασιζόμαστε στην προστιθέμενη αξία της υψηλής ταχύτητας, τα κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Μπορούμε να κερδίσουμε μερίδια της αγοράς εναντί των αερομεταφορών. Ένα παράδειγμα, σήμερα στο, στη γραμμή Παρίσι-Μπορντό έχουμε 60% μερίδιο της αγοράς και στόχος μας είναι να φτάσουμε 90-95% όπως συμβαίνει και με τη γραμμή Παρίσι-Λιόν όπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία, η σιδηρόδρομη συγγνώμη, έχουν ε, πάρει σχεδόν όλη την πελατεία στον άξονα αυτό. Καταργήθηκαν μάλιστα οι αεροπορικές γραμμές που συνέδεν το Παρίσι με τη Λιόν, διότι δεν υπάρχουν πλέον πελάτες. Ευχαριστώ, τελειώσαμε με, την παρουσία, με τις παρουσιάσεις. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ρωτώ αν οι συγγητές θέλουν το λόγο. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τις παρουσιάσεις τους. Θέλω να ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπαζέρ μας είπε ότι τα κονδύλια τα οποία βρίσκονται σήμερα στην αγορά προέρχονται από ε, ασφάλειες ή συνταξιοδοτικά ταμεία. Τι όγκος είναι αυτός, ποιο είναι το μέγεθος στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται ε, για να, ότι δεν είμαστε δηλαδή στο, στη σφαίρα του αφηρημένου. Να μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει μια αγορά με ενδιαφέρον. Στον κυρίο Χάλτερ μίλησε στην εισήγησή του γιατί εκπροσωπεί τις μεγάλες ε, εταιρείες ηλεκτρισμού. Αλλά εμείς ε, σήμερα έχουμε τις νέες υποδομές για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας υδρογόνο για την ε, μεταφορά, το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μιλάμε για την απανθρακοποίηση. Ε, χρειάζονται εδώ ε, άμεσα υποδομές και εναλλακτικέ λύσεις. Ρωτώ, εντάσσεται αυτό μέσα στο σκεπτικό της Ένωσής του, διότι μας είπε ότι άμα δεν είναι κάτι εμπορικό, δεν χρειάζεται επιδότηση. Αλλά εμείς έχουμε μία αγορά που μεγαλώνει. Θα πρέπει να θέσουμε στην υπηρεσία του πελάτη τις υποδομές. Και στον κύριο Γκιάβας θα μπορούσε να μας κάνει μία αξιολόγηση για το κάθε δημόσιο ευρώ στις, ε, για τους δύο τύπους συνεργασίας. Ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής ε, στις δύο φόρμουλες και αν υπάρχει αξία χρόνου. Δηλαδή η συνεργασία ή η εκχώρηση βελτίωσαν το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των υποδομών. Είναι πιο χρονοβόρα η προετοιμασία αυτών των, αυτών των συμβολέων ή είναι κάτι που προχωράει γρήγορα και μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος ο κύριος Άρκετ. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μάγερ που είναι πιστωτής το εξής. Υπάρχει νομίζω ένα θέμα κατανόησης μεταξύ των διαχειριστών των δικτύων και των χρηματοπιστωτών και χρηματοπιστωτριών. Θα ήθελα μια αποσαφήνιση λοιπόν για την σαφήνεια των προγραμμάτων υποδομών ιδίως που πολλές φορές οι αγορές δεν τα καταλαβαίνουν καλά και γι' αυτό δεν τους έχουν εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή να ξέρουμε και το πώς και το γιατί και τα πάντα. Και το άλλο είναι πώς υπολογίζουμε το απαραίτητο ποσοστό δημοσίου χρήματος που θα διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα για να φτάσουμε σε εμπιστοσύνη των ιδιωτών. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά ποιος τελικά ή πώς ένα συντονιστικό όργανο καταφέρνει και να περιγράψει σωστά στους διάφορους παράγοντες τα στοιχεία του προγράμματος και το ακριβές μείγμα δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Είτε μιλάμε για ομόλογα είτε για πιο κλασικούς μηχανισμούς. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από τον κύριο Κιγάρτ το εξής η συμμετοχή τελικά και η ελκυστικότητα για τους ιδιώτες εξαρτάται από το κατά πόσον είναι αποδοτικό ένα πρόγραμμα δηλαδή το κατά κάποιον τρόπο ενίκιο που καταβάλουν για να το πω έτσι υπολογίζεται φαντάζομαι σε μια αποδοτικότητα ανώτερη από την μέση. Και άρα, ξανάρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση, συνδέομαι, πώς αποτιμούμε την αποδοτικότητα ενός προγράμματος υποδομών εφόσον οι δημόσιοι παράγοντες κάνουν την αποτίμηση αυτή και προτείνουν μετά ένα είδος ενοικίασης ενώ οι ιδιώτες θεωρούν ότι είναι κερδοφόρο μόνο ότι πάει καλύτερα από το μέσο όρο. Και ερχόμαστε λοιπόν στα ίδια. Οι αγορές συμμετέχουν στις δημόσιες επενδύσεις αλλά με βάση την αποτίμηση της αποδοτικότητάς τους. Θεωρείτε λοιπόν, και τελειώνω και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος να γίνει μία αποτίμηση της αποδοτικότητας των προγραμμάτων υποδομών. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ο κυρία Βαλέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Πολύ σύντομα κύριε. Η ερώτηση είναι προς εμάς. Αυτό νομίζετε ότι θα είναι λειτουργικό, θα λειτουργήσει καλά. Διότι συχνά α, λέγεται ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν πάνε υποχρεωτικά εκεί όπου υπάρχει, υπάρχουν δημόσια κονδύλια, κρατικά κονδύλια όταν εμπλέκονται αυτά. Δεύτερον, ως επιχείρημα, τι γίνεται, θα υπάρχει κίνδυνος που θα καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα είναι ένα μέσο αυτό μόχλευσης που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί όσον αφορά ιδιωτικούς επενδυτές για την χρηματοδότηση υποδομών και τρίτων. Αν υπάρχουν δύο εταιρείες που εμπλέκονται σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, Πώς θα λειτουργήσει για αυτές τις επιχειρήσεις αυτό. Θα υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ή θα είναι ένα κοινό πλαίσιο και τα ομόλογα θα λειτουργήσουν για εκείνο το τμήμα το οποίο θα αφορά τις δικές τους δραστηριότητες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι σαφές ε, σε σχέση με την πείρα μου. Και δεύτερον, σύντομη ερώτηση προς εμάς κύριε. Εσείς κάνετε λόγο για προτεραιότητες αν όμως αυτός ο πίνακας, ο κατάλογος, θα αναφέρει προγράμματα κοινού συμφέροντος, κοινού ενδιαφέροντος, αυτό θα είναι σημαντικό για όλους, και για τα εμπορικά και για τα μη εμπορικά σχέδια. Αν είναι ένα εμπορικό σχέδιο, ίσως θα ήταν πιο δύσκολο αν δεν έχει εγγραφεί σε ένα τέτοιο κατάλογο να εξευρεθεί χρηματοδότηση από την αγορά γι' αυτό. Δεν νομίζετε ότι οι προτεραιότητες αν ενταθούν με αυτόν τον τρόπο θα επηρεάσουν τελικά την αγορά αυτών των επενδύσεων και θα δημιουργήσουν, ας το πω έτσι, ένα θέμα προ, ε, ανταγωνισμού σε σχέση με τις εταιρείες που θα επενδύουν σε αυτή την αγορά. Το αν θα είναι κανείς πάνω-πάνω στην προτεραιότητα ή πιο κάτω, αυτό θα επηρεάζει τα κονδύλια που θα διατίθενται. Έτσι δεν είναι ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τους εισηγητές οι σκιώδεις εισηγητές έχουμε 18 λεπτά στη διάθεσή μας 10 για ερωτήσεις 2,5 λεπτά στον καθένα μετά για τις απαντήσεις ο συνάδελφος Καντσά δύσκολο πρόεδρε σε ένα λεπτό με αυτά τα εξαιρετικά θέματα τα οποία έχουμε προσυζήτηση. Άρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέσσερι ε, θεωρήσει για ορισμένα σημεία. Εμείς χρειαζόμαστε σαφή σχέδια. Το business plan πρέπει να είναι σαφέστατο και για την επένδυση και για, την... και για τα κέρδη. Δεν θα πρέπει να χαρίζουμε λεφτά. Και αναφέρομαι εδώ με τα recovery plan όπου σε ελάχιστο χρόνο εμείς μοιράσαμε 4 δις, χωρίς να ξέρουμε τι ωφέλη επέστρεψαν, πρέπει να ορθολογικοποιήσουμε το σχήμα χρηματοδότησης. Αν δούμε την τσέρφα έχουμε εμείς 50 δις, όπου 50 εκατομμύρια έρχονται από την ΦΕΣΡ και από τα 40 στο τέλος του προϋπολογισμού θα μείνουν 25. Το PPP λοιπόν είναι υποχρεωτικό για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το 1,5 δις ευρώ που έχουμε προγραμματίσει σε επενδύσει. Εγώ για τα συμβόλαια είμαι υπέρ της εκχώρησης, διότι ο κίνδυνος του κυκλοφοριακού φόρτου παραμένει στο τα χέρια του δικιού του. Και μετά τι είναι τα project bond. Πρέπει να είμαστε σαφέστατοι γύρω από αυτό. Ο κύριος Μπάγκερν το ανέφερε. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει αυτό το ποιοτικό άλμα η ίδια μπαίνοντας μέσα στη χρηματοπιστωτική αγορά. Αυτό είναι το ποιοτικό άλμα που χρειαζόμαστε σήμερα. Η συνάδελφος Κούκοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι επενδύσεις ε, είναι σημαντική υπόθεση. Και οι υποδομέ είναι σημαντική υπόθεση, διότι είναι ο ταχύτερο τρόπο για μα να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση. Έμεσα αυτό θα μα δώσει την δυνατότητα να παράσχουμε, να δώσουμε πρόσθετη αξία σε διάφορου τομεί, διαφορετικού τομεί. Μία ερώτηση θα είχα προ τον κύριο Γκέρβατ. Τι γίνεται εδώ. Μας καταδείξατε ποια είναι η πείρα σας και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι που αφορά την διατήρηση, τη συντήρηση. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για την συντήρηση. Είπατε οι ίδιοι υπάροχοι θα είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση. Για ποια περίοδο, 30 ετών, 50 ετών. Και μια άλλη ερώτηση προς εμάς κύριε. Αναφέρατε τον τομέα των ενεργειακών θεμάτων, της ενέργειας. Θα ήθελα να γνωρίζω τα ορυκτά καύσιμα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι επιλέξιμα για 9 δίσσα Η κυρία Herzog, παρακαλώ. Κύριε ευχαριστώ πρόεδρε. Φαίνονται όλα εξαιρετικά θεωρητικά σε αυτό το πλαίσιο, όμως πολύ συγκεκριμένα θα ήθελα να ρωτήσω πόσο πιθανό, πιθανό είναι ότι πραγματικά θα γίνουν όλα αυτά όπως τα φανταζόμαστε εμείς εδώ. Σύντομα θα ήθελα να αναφέρω σε περιόδους όπου υπάρχει πίεση για τον προϋπολογισμό και την εξυγίανση των δημοσιονομικών και υπάρχει και δημόσια πολιτική πίεση, δεν μπορώ να κατανοήσω και να δω πώς θα ανταποκριθούμε και και τι θα κάνουμε. Κυρίως πρόκειται για το θέμα που θέλω να θέσω σε ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο τμήμα, ποιο τμήμα θα έχουν οι δημόσιες και ιδιωτικές συμπράξεις μέσα στον πυρήνα των κύριων προτεραιοτήτων προγραμμάτων και σχεδίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποια πείρα έχουμε συλλέξει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, η υπηρεσία TEN των ευρωπαϊκών διαδικτυώσεων, των ευρωπαϊκών δικτύων. Πρέπει να υποθέσουμε και να πούμε ότι θα είναι πολύ δυσχερές εγχείρημα αυτό. Διότι υπάρχει ανταγωνισμό εδώ και θέμα αρμοδιοτήτων. Αν τα είδα καλά, έχουμε ένα κέντρο πραγματογνωμοσύνης ε, ε, ε, και πρόκειται και για την πραγματογνωμοσύνη για την υποστήριξη των επενδύσεων Μέχρι σήμερα είναι δημόσιες αρχές και οργανισμοί. Τι θα κάνουμε με τους ιδιώτες, πώς θα εμπλακούν οι ιδιώτες, που ένα μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων θα πρέπει να υπομισθούν. Δεν είναι όλα αυτά απόλυτα κατανοητά. Ακούγονται εξαιρετικά και χαίρομαι αν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όλα έτσι. Αλλά με ποιο συγκεκριμένο τρόπο μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Grazie, il collega Weber. Βέμπερ παρακαλώ στη συνέχεια. Σε, ένα λεπτό. Είναι εφικτό αλλά καταπληστικό. Στον κύριο Έλντιαν. Είπατε ότι 9,1 δις ευρωπαϊκών κονδυλίων για τα 50 δις που έχουν προβλεφθεί για, συνολικά για όλο τον ενεργειακό μηχανισμό ε, της, ε, στην Ευρώπη, εντάξει σας βολεύει, αλλά για να ξεκι... εσάς προσωπικά, αλλά για να ξεκινήσει αυτό το ενεργειακό ε, δίκτυο είναι λίγο και έως ανεπαρκές. Εσείς κατα... πόσο αξιολογείτε, ποιο ποσό θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο. Στον κύριο Γκιβάρς, 37 δις Α, 31,7 διορθώνει το της. Ε, προορίζονται ως ε, καταρχήν κεφάλαιο για, την, ε, για, για να προσελκύσουν τους επενδυτές στους σιδηροδρόμους. Μας λένε ότι το 1 εκατομμύριο που επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνεπάγεται αντίστοιχα 5 εκατομμύρια κρατικά και 25 ε, ιδιωτικά στον, ε, ως επένδυση στον σιδηροδρομικό τομέα. Ο κύριος Ντεγκράντες. Όχι. Δεν θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Κράμερ. Ναι, έχουμε πείρα και έχουμε εμπειρίες σχετικά. Έχουμε εμπειρίες με τις ε, δημόσιες ιδιωτικές συμπράξεις ε, ως πρωτοβουλίες. Και όταν τα είχα παρουσιάσει στην Ελβετία, και ρώτησα ποια είναι η αντιμετώπιση τους, μου είπαν ναι, όταν είναι υπερβολικά μεγάλος κίνδυνος δεν έχουμε ιδιώτες επενδυτές. Αν αξίζει η επένδυση τότε την κάνουμε μόνοι μας εμείς οι ίδιοι. Αυτό είναι το κέριο θέμα. Έχουμε ε, πείρα και με το Channel Tunnel πώς χρηματοδοτήθηκε. Έχουμε και στο Βερολίνο ένα νέο αεροδρόμιο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αρχικά οι ιδιώτες έπρεπε να, ε, συμμεριστούν αυτές τις επενδύσεις. Έθεσαν όμως ε, τέτοιες προϋποθέσεις ε, είπαν εντάξει το, τα κονδύλια πρέπει να διασφαλιστούν όμως οι κίνδυνοι θα είναι θέματα που θα υπομίζεται το κράτος και γι' αυτό ε, όπως είπαμε αν είναι κάτι κερδοφόρο τότε το κάνει το κράτος μόνο, μόνο του μέσω των ε, ε, πιστώσεων. Πείτε μας τι γίνεται σε σχέση με αυτά τα προγράμματα που αξίζει μια τέτοια πρωτοβουλία από πλευράς του δημοσίου όχι μόνο για τους ιδιώτες θα μας ενδιέφερε αυτό. Grazie, σας ευχαριστώ. Και εγώ θα είχα μία ερώτηση προς τον κύριο Χάλντεν ως εκπρόσωπο ρυθμιστικών αρχών. Πιστεύετε ότι καλό θα ήταν να υπάρξουν επενδύσεις ε, όσον αφορά τον δημόσιο τομέα στον, στις υποδομές ε, για το φυσικό αέριο. Από την άλλη πλευρά οι υποδομές για το φυσικό αέριο είναι ένα είδος μονοπωλίου και μέσα στο τρίτο πακέτο για την ενέργεια τι θα γίνει σε σχέση με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για κάποιες χώρες. Αυτό θα αύξενε τα κέρδη των μονοπωλίων, του μονοπωλιακού κεφαλαίου και θα υπήρχαν ίσως και προβλήματα άλλοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις υποδομές. Επόμενη ερώτηση ερώτηση προς τον άλλο ομιλητή για τα project bonds, τα ομόλογα έργου. Τι γίνεται με τις χώρες χαμηλού κινδύνου. Θα ήταν ασφαλές να λειτουργήσουν τέτοιες δράσεις για τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε δέκα χρόνια πού θα βρισκόμαστε. Μπορεί ίσως να βρούμε ότι τα ομόλογα έργου χρησιμοποιούνται μόνο σε τέτοιες χώρες. Ευχαριστώ. κύριος Πίρκερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να μου απαντήσει αυτό το ερώτημά μου όμως παρόλα αυτά θα το διατυπώσω. Πρόκειται για την υπέρβαση αντιστάσεων όσον αφορά την, ε, ε, τα έργα υποδομής. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει θετική επίπτωση στην οικονομία από τέτοιες υποδομές σε σχέση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα για παράδειγμα. Ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της ε, διεύρυνσης των δικτύων υψηλής απόδοσης. Από την άλλη πλευρά και για την πείρα μας υπάρχει και ηχητική επιβάρυνση και όχλη και γι' αυτό εξειδικευμένα προγράμματα αντιμετωπίζουν αντιστάσεις και διαφωνίες. Μπορεί να είναι και θέματα τουρισμού ή ε, διαμαρτυρίας πολιτών λόγω τέτοιων προβλημάτων. Ερώτησή μου, υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια εμπειρία, υπάρχει κάποια εμπειρία πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα και τέτοιες ε, αντιδράσεις. Υπάρχει προγραμματισμός και σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με ε, το υλικό που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς για παράδειγμα με την, τον ανασχεδιασμό τέτοιων διαδρομών με την διάνοιξη σειράγκων ε, ε, όσον αφορά τούνελ για παράδειγμα στις διαδρομές υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται ώστε να ανταποκριθούν στις ευαισθησίες των περιοίκων. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Επειδή πιέζει πολύ ο χρόνος, κάποιες σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, πώς αντιδρούν ε, οι ιδιώτες επενδυτές ε, στο κόστος που αυξάνεται παντού κατά τη διάρκεια των ε, εκτελέσεων των έργων ενός ε, σχεδίου ε, αυτοκινητοδρόμου, π.χ. σιδηροδρομικών γραμμών κτλ. Πώς αντιδρούν σε σχέση με την αύξηση του κόστους. Πώς τέτοια κριτήρια μπορούν, για παράδειγμα, σε σχέση με την ολοκλήρωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων να εντάσσονται σε τέτοιου είδους σφαιρικές δραστηριότητες. Τρίτη ερώτηση. Υπήρξε μια μελέτη για την ιδιωτική δημόσια σύμπραξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στο παρελθόν συντάχθηκε και διαπίστωσε ότι με τέτοια προγράμματα και σχέδια μεγάλου χρονικού ορίζοντος ε, είναι δύσκολο να είναι άμεσα κερδοφόρα τέτοια προγράμματα δράσεων δημόσιας ιδιωτικής ε, σύμπραξης. Αυτά τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης εξακολουθούν να ισχύουν ή όχι. Τι είναι υπέρ ενός μεγάλου χρονικού ορίζοντος ε, για τον κερδοφόρο χαρακτήρα τέτοιων επενδύσεων. Τελευταία ερώτηση. Κατά πόσον είναι ιδιωτικές αυτές οι ιδιωτικές επενδύσεις. Τι γίνεται με τους θεσμικούς επενδυτές. Ε, οι δήμοι και οι κοινότητες, οι περιφέρειες θα είναι ιδιώτες εντός εισαγωγικών. Ποιοι είναι αυτοί οι ιδιώτες σε εισαγωγικά Συγκεκριμένη ερώτηση. Υπάρχουν κάποια δεδηλωμένα ενδιαφέροντα ή συμφέροντα από κάποιους ιδιωτικούς επενδυτές για τέτοια προγράμματα και σχέδια. Διότι αυτό είναι ενδιαφέρον να δούμε. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να διασφαλιστεί μια τέτοια χρηματοδότηση ή θα είναι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Η συνάδελφος Διογόν, τελευταία τοποθέτηση. Ευχαριστώ και σχεδια διοτι αυτο ειναι ενδιαφερον να δουμε υπαρχει καποια πιθανοτητα να διασφαλιστει μια τετοια χρηματοδοτηση η θα ειναι μονο σε θεωρητικο επιπεδο η τελευταια τοποθετηση ευχαριστω και συντομα Ορισμένες εμπειρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τούνελ κάτω από την ε, Μάχη, το Ίτερ ή ο Γαλιλαίος που κόστησαν δύο ή τρεις φορές πάνω από την τιμή που προαναγγέλθηκε, οδηγούν στο να έχουμε ε, ερωτήσεις σήμερα για το κατόφλι απόδοσης. Σήμερα βέβαια οι νέοι κανόνες μας υποχρεώνουν να αναζητήσουμε μορφές συνεργασίας και να διευκρινίσω την ερώτηση του κυρίου Ρικέ. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι σχετικές τιμές κατοφλίου, δηλαδή δημόσιας χρηματοδότησης και διάρκειας του σχεδίου, όπου εγγυόμεθα ότι δεν ιδιωτικοποιούμε μόνο τις ε, ε, απώλειες, αλλά δεν κρατικοποιούμε ειδικά το, το, ρίσκο. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να εγγυθούμε ότι το δημόσιο χρήμα εγγυάται, ε, ε, είναι εγγυμένο από την επένδυση του ιδιωτικού τομέα και πώς το νίκη αυτό πληρώνει το χρέος αλλά και αποδίδει. Εδώ έχω καμιά δεκαριά ερωτήσεις και 25 δευτερόλεπτα για την κάθε μία να δώσω. Λοιπόν, αρχίσω από την αρχή. Αν θέλει κανείς θα συνεχίσουμε μετά ιδιαίτερος. Λοιπόν, 95 με 7 υπήρξαν 300 δοσοληψίες με τέτοια ομόλογα έργου για υποδομές. Η αγορά είναι πολύ μεγάλη όντως και ο τομέας των υποδομών ιδιαίτερα. Ιδίως πριν την κρίση βέβαια. Κάποιος άλλος με ρώτησε για τους τρόπους αποσαφήνισης των σχέσεων του χρηματοδότη με τον χρηματοδοτούμενο. Αυτό γίνεται από την ΕΤΕ. Αυτός είναι ο σκοπός της ακριβώς. Δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία από την πλευρά των επενδυτών, άρα πρέπει τέτοια όργανα να φροντίζουν την οργάνωση και υποδομή της εκτέλεσης των ομολόγων. Οι διαχειριστές των δικτύων είναι εκείνοι που χορηγούν τις πληροφορίες στις τράπεζες. Άλλο ερώτημα. Να δω γιατί μου διαφεύγει. Ποιοι ακριβώς είναι οι επενδυτές και οι επενδύτριες, οι θεσμικοί, οι ιδιώτες. Είναι πολλοί και διάφοροι. Υπάρχουν τεράστιοι αριθμοί συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστικών εταιριών που επενδύουν. και με ιδιωτικά ομόλογα γιατί είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδου επενδύσει και αναλήψει κινδύνου. Αυτό που δεν, στο οποίο δεν είναι συνηθισμένοι είναι τα κρατικά ή τα ομόλογα έργο. Σε όλα τα σχέδια που συζητούμε σήμερα, τα περισσότερα μάλλον δεν είναι τύπου πι. Another question is, do I think it's going to work? Can't remember. Σύμπραξης δηλαδή δημοσίων και ιδιωτών. Εγώ έχω 33 ετή εμπειρία και σε πολλούς τομείς της αγοράς καθώς και στην εταιρεία ο τείχος του Αδριανού και στην ΕΤΕ. Τέτοιες δομές υπάρχουν για εδώ και πολλά χρόνια και δεκαετίες και δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Ε, πώς υπολογίζουμε τη συμμετοχή δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Στον τομέα του PPP δεν υπάρχει τεράστια χρηματοδότηση. Το θέμα είναι πώς ακριβώς διευθετείται η συμφωνία, ποιες είναι οι ευθύνες των κυβερνήσεων όταν λάβουν τα χρήματα. Όταν οικοδομηθεί το έργο περατωθεί και δοθεί στην κυβέρνηση χρειάζεται κάποιο ενίκιο για 20-25 χρόνια. Τώρα ο λόγος, η κατανομή δεν θα σκεφτόμαστε έτσι εμείς τον λόγο δηλαδή δημοσίων με ιδιωτικών επενδύσεων. Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Τελεία. Αυτά, μάλιστα. Μα έχουμε και άλλο γύρο γι' αυτό. Μετά, άμα θέλετε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ξαναλέτε κι άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήματα μου τέθηκαν. Το ένα αφορούσε τις νέες υποδομές για ενεργειακές πηγές και αν αυτό το σκέφτονται ή το γνωρίζουν οι ρυθμιστές και οι ρυθμίστριες και αν ισχύει και για τα ορυκτά καύσιμα εδώ μιλάμε για επενδύσεις σε υποδομές δικτύωσης, δηλαδή υποδομές σύνδεσης των διαφόρων τμήματων της Ευρώπης με νέες πηγές. Οι ρυθμιστές και οι ρυθμίστριες νομίζω τα γνωρίζουν αυτά, αφού ενθαρρύνουν τέτοιου είδους επενδύσεις, ας πούμε στις ανανεώσιμες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να γίνουν εκεί σε αυτό το τομέα επενδύσεις στις υποδομές τους. Στα λεγόμενα έξυπνα δίκτυα το ίδιο ισχύει. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να διαδοθούν καλύτερα οι βέλτιστες πρακτικές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ευρωπαϊκή υπηρεσία που στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Η απάντηση λοιπόν είναι ναι, το γνωρίζουν. Βέβαια ο τομέας αυτός αλλάζει συνεχώς. Άλλο θέμα ήταν οι προτεραιότητες. Αν κάτι έχει υψηλή προτεραιότητα δεν σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθεί και ευκολότερα. Δείχνει απλώς ότι είναι πιο επίγονο χαρακτήρας του για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ευρώπης. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης εξαρτώνται από παράγοντες όπως το αν το σχέδιο αυτοχρηματοδοτείται, αν είναι οικονομικά σταθερό και αν πόσο κίνδυνο εμπεριέχει κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει μεν κάποια σχέση με το, τη θέση του προγράμματος στις προτεραιότητες αλλά δεν ακολουθεί ότι η υψηλότερη προτεραιότητα είναι καλύτερη ή ευκολότερη χρηματοδότηση. ...9,1 δισεκατομμύρια δεν αρκούν. Δεν είχα πει αυτό όμως. 9,1 δισεκατομμύρια είναι κάτι χρήσιμο αλλά όχι ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση με τις συνολικές επενδύσεις που απαιτούνται. Χρειάζεται λοιπόν να εξαρτώμαστε ακόμη και από ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης. Οι εταιρείε δικτύωσης όταν παίρνουν χρήματα από τις αγορές για να επενδύσουν πρέπει να έχουν μια πιο απλοποιημένη διαδικασία. Το 9,1 δισεκατομμύρια άμεσης χρηματοδότησης πρέπει να δοθεί. Είναι απαραίτητο αλλά δεν αρκεί ούτε μπορεί να χρηματοδοτηθεί με τον συνήθι τρόπο. Εγώ δεν έχω καμιά άποψη ως προς το κατά πόσον το 9,1 δισεκατομμύρια στερλινών αρκεί όχι, κανείς μάλλον δεν ξέρει. Θα το δούμε. Καλά, ας σταματήσω, εντάξει. Ε. Ευχαριστούμε. Και τώρα τελευταίος το Τβάρετ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τέσσερα μόνο θέματα που τέθηκαν γιατί αλλιώς δεν αρκεί ο χρόνος. Για τη διάρκεια των συμβολέων 15 περίπου χρόνια και για ορισμένα 25, όσο για το Turbo Do 50 χρόνια. Δεύτερον, οι πολλαπλασιαστικές ή μη επιπτώσεις του χρονοδιαγράμματος. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα γιατί η διάρθρωση των σιδηροδρομικών προγραμμάτων, η κατάστρωση τους χρειάστηκε πολύς χρόνος Βέβαια η δημιουργία ενός προγράμματος είναι σχεδόν 10.000 έγγραφα. Χρειάζεται πολύ χρόνος λοιπόν και μέχρι τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν και ιδιαίτερα γρήγοροι, αλλά μπορέσαμε τουλάχιστον να ταυτίσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες και μπορούμε τώρα να δούμε πού μπορεί να υπάρξει επιτάχυνση στο χρονοδιάγραμμα το ότι χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι σημαίνει ότι είναι κάτι καινούριο και μπόρεσαν να οικοδομηθούν δύο γραμμές υψηλής ταχύτητας ταυτόχρονα χάρη στο ΠΠΠ. Δηλαδή, μία γραμμή οικοδομήθηκε ως συνήθως με τις δημόσιες προμήθειες και τρεις άλλες αποκλειστικά με ΠΠΠ. Υπάρχει κανονική δημόσια χρηματοδότηση με ισχυρή εισφορά του κράτους κατά 75% και το υπόλοιπο 25% δεν είναι δημόσια επιχορήγηση γιατί προκύπτει από τα έσοδα της δημόσιας εταιρείας. Στις υπόλοιπες όμως τρεις γραμμές ήταν πολύ χαμηλότερη η κρατική επιχορήγηση. Τώρα για την αποδοτικότητα και ελκυστικότητα. Υπάρχουν ορισμένα λεπτά θέματα όπως η αύξηση του κόστου σε σχέση με τις προβλέψεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου εκτός από τους κινδύνους που δεν αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας οι υπόλοιποι κίνδυνοι συνήθως αναλαμβάνονται από τους ιδιώτες. Όταν βέβαια χρειάζεται 6-6,5 χρόνια για την πραγματοποίηση ενός μιας υποδομής, εφαρμόζεται μία καταποκοπήν πληρωμή μέχρι τη λήξη του συμβολέου. Ο κατασκευαστής δεν έρχεται να μας ξαναπεί θέλω κι άλλα. Σήμερα θεωρούμε ότι ο ιδιωτικό τομέα ανέλαβε ιδιαίτερα ψηλούς κινδύνους και αναμένουμε βελτιώσεις ως προς την σύλληψη των προγραμμάτων και την εκτέλεσή τους. Δεν είμαι μεν μηχανικός, αλλά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Ας πούμε, στις γραμμές που γίνονται πάνω σε μπετόν. Αναμένουμε τις βελτιώσεις αυτές, αν και δεν έχουμε ακόμη όλα τα στοιχεία. Και τελειώνω με κάτι με το εξής δυνατότητα να εφαρμοστεί με λανθασμένο τρόπο κάποιο σχέδιο συντονισμού ιδιωτικού, συγχρηματοδότηση ιδιωτικού με δημόσιο τομέα είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δίνω το λόγο και την Προεδρία στον Μπράιαν Σίμψον, πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών. Για το δεύτερο πάνελ έχουμε ένα τέταρτο καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουν τώρα κάποιοι θέσεις. Θα χρειαστούν και άλλα πρόσθετα πέντε λεπτά. Okay, let's try and get started. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε λοιπόν πάλι. Λιγότερα από 45 λεπτά για αυτό το δεύτερο πάνελ. Θα είμαι ανελέητος. Ανελέητος είναι ο όρος που έρχεται στο νου μου με τρεις αγορητές. Δεν θα κάνω όλη την εισαγωγή, διότι αυτό θα πάρει και άλλα δύο λεπτά. Θα περάσω αμέσως στον κύριο Κόμακ Μορφή Διευθυντή Δράσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχετε τον λόγο κύριε. Κάθε αγορητή θα έχει 10 λεπτά και μετά θα αποφασίζω τι θα γίνεται σε σχέση με τις ερωτήσεις, με τα αιτήματα τα οποία θα έχουμε ανάλογα με τους αγορητές. Έχετε τον λόγο κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Θα μιλήσω εξ ονόματο τη ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μετά από τι προηγούμενε παρεμβάσει που κάλυπταν το ίδιο ως θέμα ουσία, αλλά και τι προοπτικές τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με προοπτική όσον αφορά τα μέσα για την χρηματοδότηση των υποδομών, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον ρόλο τη ιδιωτική ε, επένδυση των ιδιωτών, των ε, συμπράξεων ιδιωτών και δημοσίου και την δυνατότητα να μπορέσουν με τέτοια μέσα και ομόλογα να προχωρήσουν αυτά τα έργα από τις επενδύσεις. Λοιπόν. Okay. Okay, excuse me. Sorry. Mr. in particular has mentioned... Ιδιαίτερα αναφέρθηκε πιο πριν, αναφέρθηκαν τα θέματα τα οποία αφορούν τη χρηματοδότηση των υποδομών από πλευρά του δημοσίου και όσον αφορά παράγοντες και συντελεστές που συγκλίνουν. Ένας είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα των ε, ασφαλιστικών εταιριών που έχουν εξαφανιστεί ως ε, δυνατότητα ε, διασφάλισης τέτοιων κινδύνων όσον αφορά τις δημόσιες υποδομές. Δεύτερον, η απομόχλευση σε μεγάλο βαθμό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή τεκταίνεται ιδιαίτερα στις τραπεζικές αγορές και ιδιαίτερα όσο αφορά τις απαιτήσει που αυξάνουν το κόστος μακροπρόθεσμα, το μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό κόστος. Και κάτι άλλο φυσικά είναι και η χρηματοοικονομική κρίση. η περιορισμοί όσον αφορά τα κονδύλια από πλευρά δημόσιων ε, προϋπολογισμών, κρατικών προϋπολογισμών. Υπάρχει η ανάγκη σε μεγάλο βαθμό επενδύσεων. Οι υποδομές είναι η κοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αναγκαίο στοιχείο για την ανάπτυξη. Αναγκαίο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ανάλογα με τα μεγέθη που κάνουμε λόγο, κάνουμε λόγο για ένα 3 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Πολύ μεγάλη ανάγκη η οικονομική αυτή. Ερώτημα, πώς θα καλυφθεί αυτή η ανάγκη Πώς θα υπάρξει μόχλευση με την χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα πρέπει ο ιδιωτικός τομέας, οι ιδιώτες επενδυτές να εμπλακούν σε αυτό το μακροπρόθεσμο εγχείρημα και να αντιμετωπιστούν θέματα όπως αφορά και την δημόσια υπερχρέωση όσον αφορά την δυνατότητα διασφάλισης κονδυλίων για αυτές τις υποδομέ. οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δράει εδώ και 50 χρόνια και η κύρια υποδομή είναι, η κύρια, το κύριο έργο είναι υποδομέ από πλευρά τη. Χρηματοδοτήσαμε προγράμματα και σχέδια παντού στην Ευρώπη τι τελευταίε δεκαετίε από μια δομή που ήταν πιο παραδοσιακή πιστώσεων και δανείων στι κυβερνήσει, λαμβάνοντα υπόψη και βοηθώντα την ανάπτυξη νέων αγορών, παράδειγμα τη ιδιωτική και δημόσια σύμπραξη, PPP,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 Partnership. Αυτό έχει συγκεκριμένες ανάγκες. PPP χρηματοδότηση για το project, για το έργο που πρέπει να επιτελεστεί, για παράδειγμα όσον αφορά τον αδιούχο πάροχο. Έχουμε νέα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται τα τελευταία ε, χρόνια. Για παράδειγμα με χαμηλά επιτόκια δάνεια και ε, να ε, παρασχεθεί αρρωγή και υποστήριξη. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα στις μεταφορές ε, και τα διάφορα άλλα πιστοτικά μέσα τα οποία επιτρέπουν την κάλυψη χρηματοοικονομικών κινδύνων όσον αφορά τις συναλλαγές αυτές ε, και τα φαινόμενα και περιπτώσεις κινδύνων όσον αφορά τις, ε, τους παρόχους. Ε, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έδινε και δυνατότητα μέσω ομολόγων για τη χρηματοδότηση ε, αυτών των προγραμμάτων και με την δυνατότητα δημόσιας ιδιωτικής σύμπραξης. Η ΕΤΕ, ΕΤΕΠ έχει αποκτήσει όλο και σημαντικότερη, μεγαλύτερη σπουδαιότητα σε σχέση με την χρηματοοικονομική κρίση. Βλέπετε κάποια μείωση που σημειώνεται το προηγούμενο έτος μειώσαμε τις δραστηριότητες μας από το πολύ υψηλό επίπεδο αλλά πάλι σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με ευθυγράμμιση με το μέσο που χρησιμοποιούμε. Όμως ο επιμερισμός των ε, σχεδίων ε, σημειώνει μεγάλη άνθηση και αυτό έχει σημασία κλειδιού. Είναι μεγάλη σπουδαιότητα η συνέχιση των προγραμμάτων αυτών ακόμα και σε ε, περιόδους αντικσοτήτων όπως η σημερινή συγκυρία. Τα TENS, τα διευρωπαϊκά δίκτυα έχουν μεγάλη σημασία στις δραστηριότητες μας. Εδώ μπορείτε στο γράφημα αυτό να δείτε το υψηλό επίπεδο προτεραιότητα σε σχέση με τις πιστώσεις και τα δάνεια δάνεια που χορηγούνται από την ΕΤΕΠ σε σχέση με την οικονομική κρίση και να δείτε και τη σημασία, τη σπουδαιότητα αυτών των δράσεων. Βλέποντας τα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες ξεκινήσαμε από χαμηλά επίπεδα και στα πρώτα χρόνια ιδιαίτερα στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυξήθηκαν όμως αυτές οι δράσεις και επεκτάθηκαν και σε διάφορες άλλες χώρες όπου τώρα έχουμε σημαντική εξάρτηση στις ε, αγορές αυτές ε, στην Ευρώπη μέσω αυτών των μέσων. Ανέφερα και την περίοδο κρίσεως και τις πιστοτικές δράσεις της τράπεζας και την ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών μέσων. Ιδιαίτερα εδώ θέλω να τονίσω την διασύνδεση της Ευρώπης, Interconnecting Europe και το LGTT Instrument και όσον αφορά την δανειοδότηση, τα, ε, η πρωτοβουλία ε, ομολόγων έργου, Project Bonds, έχει αναλυφθεί και υπό ε, την προοπτική έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο του επόμενου μήνε για να αναπτυχθεί στο πλήρες, στον πλήρη βαθμό μέχρι το 2014-2020 και την χρήση αυτού του μέσου σε αυτή την προγραμματική περίοδο με το Interconnecting Europe Facility, το μέσο για τη διασύνδεση τη Ευρώπη με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Επίση, για τι υποδομέ, ιδιαίτερα όσον αφορά το δημόσιο, τι κρατικέ αρχέ και την ευρωπαϊκή, ε, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημόσιας Ιδιωτικής Σύμπραξης για την ανταλλαγή εμπειρίας και ε, πείρας, ώστε να υπάρξει όφελος από τις ανταλλαγές αυτές και τις ε, τη διασπορά της, ε, των πληροφοριών. Το Project Bond, το, το ομόλογο έργο είναι ένα μέσο για να μπορέσει να δώσει δραστηριότητα σε κινδύνους που θα βρίσκονται κάτω από το ανώτατο επίπεδο. Αυτό διευρύνει την ποιότητα, επεκτείνει την ποιότητα του κεκτημένου για τους παρόχους δανείων. Υπάρχουν άλλοι senior debt holders ε, έναντι των ε, subordinated debt holders. Υπάρχει μικρότερη θα έλεγα έκθεση όσον αφορά τους κινδύνους για τέτοιου είδους έργα. Η πρόθεση αυτού, αυτής της δομής είναι να παράσχουμε υποστήριξη και να ενθαρρύνουμε τις κεφαλαιακές αγορές να δράσουν και να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα υποδομών. Αυτό είναι και ένας τρόπος να υπάρξει μόχλευση από πλευράς κεφαλαίων, ώστε τα κονδύλια τα οποία θα δεσμεύονται από πλευράς του προϋπολογισμού του Ευρω... του... της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πολλαπλή, πολλαπλό αντίκτυπο όσον αφορά την πραγματική τους δράση. Τελικά είναι ένας τρόπος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μπορεί να κάνει περισσότερα και είναι ένας τρόπος να δώσει πρόσθετη μόχλευση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιπρόσθετα στην πραγματοποίηση και στην παροχή υποστήριξης για τέτοιου είδους ε, ε, εκτέλεση έργων υποδομών. Η συνεισφορά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας ε, είναι συγκεκριμένη με ανώτατα κονδύλια που προβλέπονται για κάθε πρόγραμμα. Αναλαμβάνουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζας την κάλυψη κινδύνων όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και βλέπουμε ότι οι δυνατότητες κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μέσου μπορεί να δώσει την δυνατότητα κονδύλια να μπορούν να χρησιμοποιούνται πολλαπλά. Τώρα για, τον πολλαπλασιαστικό, για την πολλαπλασιαστική χρήση ε, multiplier ε, κονδυλίων που παρέχονται και την μόχλευση από τα 230 εκατομμύρια που παρέχονται υπό τα διάφορα κονδύλια 10T και 10E και CIP, οι προσδοκίες ποιες είναι. Οι προσδοκίες είναι ότι τα 230 εκατομμύρια θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να παράσχει μέσα τα οποία θα οδηγήσουν στο να προσεγγίσουμε περίπου τα 700 εκατομμύρια. Τριπλάσια μόχλευση δηλαδή σε σχέση με τα 230 εκατομμύρια. Και έχοντας υπόψη τα ομόλογα αυτό θα δώσει δυνατότητα μόχλευσης 19 ή 20 φορών. 20 πλάσια μόχλευση. Αυτά όλα εξαρτώνται φυσικά από την χρήση των ομολόγων και αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο είναι εικονικής χρήσης ε, για να σας ε, καταστεί αυτό πιο κατανοητό. Θα δώσει την δυνατότητα στους ε, ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα για να επιτευχθεί μια πιστοδότηση, διασφάλιση πιστώσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι θελκτική, ελκυστική για τέτοιου είδους ιδιώτες επενδυτές. Και τέλος, ένα άλλο στοιχείο των δραστηριοτήτων της τράπεζάς μας είναι επενδύσεις με ομόλογα σε έργα υποδομών. Και αυτό είναι κάτι που είμαστε πρόθυμοι να αναπτύξουμε υπό το εγχείρημα Connecting Europe Facility και ομόλογα σε σχέση με την ε, ε, προσέγγιση κινδύνων ε, η τα ομόλογα είναι ένα σημαντικό ε, στοιχείο για το χρηματοοικονομικό μείγμα το οποίο χρησιμοποιούμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Μάρφη. Τώρα ο υπεύθυνο της Γενικής Διεύθυνσης MOVE. Ορίστε κύριε Γιάννη Ερίκο. Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ένωση είναι να βρει τρόπους επένδυσης για την ανάπτυξη. Και η επένδυση στις τρεις ε, βιομηχανίες ε, σύνδεσης είναι τρόπος ανάπτυξης της Ευρώπης. Γιατί έτσι οι οικονομίες και η κοινωνία μας γίνονται πιο ανταγωνιστικές και δίνουν μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή στην εσωτερική αγορά. Τέτοιες επενδύσεις υποστηρίζουν και το πρόγραμμά μας βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών. Επίσης πρόκειται για επενδύσεις που στηρίζουν άμεσα τις βιομηχανίες μας σύνδεσης και επικοινωνία. Πρόκειται λοιπόν και για καινοτομία και βιομηχανική πολιτική. Οι μαζικές επενδύσεις στις τρεις βιομηχανίες σύνδεσης που θα απαιτηθούν τα επόμενα 10 και 20 χρόνια είναι μια τρομερή πρόκληση. Το ΣΕΦ συμβάλλει σε αυτό το στόχο. Δεν είναι η μοναδική απάντηση στην πρόκληση αυτή, αλλά ελπίζουμε εδώ στην Κομισιόν ότι θα μπορέσει να παίξει το ΣΕΦ έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενωσιακή διάσταση των επενδύσεων αυτών. Θα έρθουν επενδύσεις και από τη βιομηχανία, από τις κεφαλαιαγορές και από τράπεζες φυσικά, ιδιαίτερα από την ΕΤΕ. Επίσης όμως και από δημόσιες πηγές εθνικές ή ενωσιακές. Η πρόκληση λοιπόν που αντιμετωπίζει το Connecting Europe είναι πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν αυτές οι επενδύσεις και πώς ένα τμήμα τους θα στοχεύθει στην ζωτικότατη ενωσιακή διάστασή τους. Λοιπόν, για να δούμε πώς μπορεί η Ένωση να διευκολύνει το Connecting Europe, χρειάζονται, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τρεις διαστάσεις. Πρώτον, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο σχεδιασμού, δεύτερον ταύτιση, καλύτερη ταύτιση του ωφέλους που θα έχουμε από την ενωσιακή διάσταση και τρίτον καλύτερος συνδυασμός δημόσιος χρηματοδότησης με άλλη. Για το σχεδιασμό η Κομισιόν μαζί με το Connecting Europe προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στις μεταφορές και αλλού που ταυτίζουν την ενωσιακή διάσταση αυτών των βιομηχανιών ε, σύνδεσης και επικοινωνιών και προτείνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, καταρχήν τα κράτη-μέλη αλλά και ενδιαφερόμενους από την βιομηχανία σε περιφερειακό επίπεδο και εκείνους που εφαρμόζουν, την, ε, που κατασκευάζουν την υποδομή, συνεργασία γενικώ. Η δέσμη ΣΕΦ λοιπόν συμπεριλαμβάνει προτάσεις για την ανάληψη δεσμεύσεων από όλους τους ενδιαφερομένους στο σχεδιασμό και στην κατάστρωση πολιτικής. Επίσης είπα χρειάζεται καλύτερα προγράμματα προτεραιότητες που θα ταυτιστούν από την Κομισιόν μέσω του Connecting Europe στην προσθήκη του οποίου αναφέρονται οι κύριες προτεραιότητες για τους τρεις τομείς που θα συμβάλλουν στην περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις και τα επόμενα 7 χρόνια θα επιτρέψουν στο Connecting Europe αλλά και σε μεγαλύτερη προγραμματική περίοδο να αναπτύξει, να ταυτίσει τυχόν ελλείμματα. Χρειάζονται επίσης καλύτερα προγράμματα μέσω καλύτερης συνεργασίας μεταξύ τους και συνδυασμού και εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πώς να ταυτιστούν προγράμματα οριζόντια Έχουμε και μερικά εργαλεία για καλύτερο συγχρονισμό και προετοιμασία των επενδύσεων σε όλα τα κράτη-μέλη. Πολλά από αυτά είναι μεμονωμένα τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, ιδιαίτερα στις μεταφορές. Ας πούμε οι διάδρομοι που συνδέουν απομακρυσμένες περιφέρειες για να υπάρξει συνδυασμός και συντονισμός και μεταξύ περιφερειών. Γίνεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια για την καλύτερη προετοιμασία των προγραμμάτων. Οι ενεργειακοί ρυθμιστές επίσης κάνουν το ίδιο όπως και στις μεταφορές και η ΕΤΕ μαζί με την Κομισιόν και τις άλλες ενωσιακές υπηρεσίες, ρυθμιστικές ή μη, θα αρχίσουν την επεξεργασία συγκεκριμένων προγραμμάτων ώστε να είναι έτοιμο το 14 το ΣΕΦ να λειτουργήσει με συγκεκριμένο κατάλογο και απαρίθμηση προγραμμάτων και σχεδίων. Τέλος, χρειάζεται καλύτερη χρηματοδότηση. Μίλησαν και οι προηγούμενοι για τη χρηματοδότηση με περισσότερη εμπειρία από μένα αλλά πρέπει παρόλα αυτά να τονίσω ότι η χρηματοδότηση είναι σημαντικό τμήμα της επένδυσης. Ιδιαίτερα, in transport and the work to be done. ιδιαίτερα στις μεταφορές, αλλά και στα προγράμματα που συζητάμε μέχρι το 2014 για το συνδυασμό με τον τραπεζικό τομέα ώστε τα κεφάλαια αυτά να μπορέσουν να διατεθούν αποτελεσματικότερα. Το ΣΕΦ υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία και την μέθοδο τους μηχανισμούς κατανομής των κινδύνων καθώς και τα περίφημα ομόλογα έριγου που θα είναι έτοιμα για μέχρι το καλοκαίρι. υπάρχει και το Ταμείο Μαργαρίτα και για το ICT που λέμε και για τις μεταφορές. Ευθύνη όμως των ίδιων των προγραμμάτων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι να συνεννοηθούν μαζί μας για την καλύτερη δυνατή χρήση των δυνατοτήτων. Έχουμε εμπειρία, υπήρξαν επιτυχίες, και ορισμένες βέβαια ε, αποτυχίες αλλά που μπορούν και αυτές να μας δώσουν μαθήματα. Για να μιλήσω πάλι για τις μεταφορές υπάρχει πολλά γνωστά προγράμματα όπως η παρουσίαση που έγινε για τον Μπουρδό και Υπάρχουν εκεί δυνατότητες χρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα καθώς και τις κεφαλαιαγορές. Το ΣΕΦ επίσης αφορά δημόσια ευρωπαϊκή ενωσιακή χρηματοδότηση και προετοιμάζοντας το Connecting Europe περάσαμε πολύ χρόνο συνεννοούμενοι με τους συναδέλφους για να δούμε πού χρειάζεται να συνεχιστεί η δημόσια επιχορήγηση και πού όχι είχαμε πει ότι θα μπορούσε η εθνική χρηματοδότηση να δίνεται από την Ένωση κατευθείαν αντί από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε η ενωσιακή χρηματοδότηση να βασίζεται σε πραγματικές ευρωπαϊκές ε, προτεραιότητες. Βέβαια δεν θα είναι το εύτο μοναδικό εργαλείο. Υπάρχουν και τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας και τα διάφορα εργαλεία για την περιφερειακή πολιτική. Το πρόβλημα κύριε Πρόεδρε είναι πώς τα προγράμματα αυτά θα τα συνδυάσουμε και το παράδειγμα του Τουρ Μπορντό δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες πολλαπλής χρηματοδότησης. Τώρα για το συνολικό ποσό των 50 δισεκατομμυρίων, το ποσό αυτό νομίζω ότι συμβαδίζει με τον κατάλογο των σχεδίων, αλλά ε, πρέπει να δούμε αν είναι σωστά προετοιμασμένα. Είναι πάντως ένα ελάχιστο ποσό και ελπίζουμε να πείσουμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διαθέσει τουλάχιστον το ποσό αυτό. Τώρα ο αντιπρόεδρος της Deutsche Telekom. Εγώ θα τηρήσω άτεγκτα το χρόνο, 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω ότι με προσκαλέσατε σε αυτή την ε, ακρόαση παρουσιάζοντας τις απόψεις μας για την ε, διασύνδεση στην Ευρώπη. Θέλω να τονίσω ότι εμείς ως ιδιώτες υποστηρίζουμε πολύ αυτές τις προτάσεις. Με μια πρώτη ματιά όσον αφορά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ατζέντας συνειδητοποιεί κανείς αμέσως ότι θέλουμε να επενδύσουμε σημαντικά στο ευρωπαϊκό ευρύ φάσμα, να έχουμε τα, τα 30 MB όσον αφορά τον πληθυσμό και να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε 50% όσον αφορά τα 400 MB ανά δευτερόλεπτο οι ε, επιχειρήσεις ε, ε, δεσμευόμαστε να τα καταφέρουμε, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας να τα καταφέρουμε. Γι' αυτό είναι οι δημόσιες επενδύσεις μεγάλη σημασία, ώστε να μπορέσουν να διασφαλίσουν κεφάλαια εκεί όπου χρειάζονται. Βλέπετε στο γράφημα ότι καθυστερούμε, έχουμε, χωλένουμε για να επιτύχουμε τους στόχους. Πολλά μπορούν να γίνουν. Δύο στοιχεία υπάρχουν σε σχέση με το μέσο διασύνδεσης της Ευρώπης, το οποίο υποστηρίζουμε το μέσο διεύρυνσης πιστώσεων ώστε να υπάρχει μόχλευση και διαχείριση μέσω ενό οργανισμού που θα διαχειρίζεται τα κονδύλια, να διασφαλίζονται οι επενδύσεις και να υπάρχουν πιστώσεις για τον ιδιωτικό τομέα. Και από την άλλη πλευρά είναι πολύ σημαντικό η πτυχή όσον αφορά τις άμεσες επιχορηγήσεις, όσον αφορά μη κερδοφόρους τομείς. Χρειαζόμαστε και τα δύο σκέλη για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε για να πετύχουμε τους στόχους της ψηφιακής ατζέντα για μια ερώτηση που ήδη διατυπώθηκε αν υπάρχουν αρκετά κονδύλια 300 δις ε, ευρώ προβλέπονται για αυτή την περίοδο είναι ένα κλάσμα όμως των συνολικών κονδυλίων που χρειάζονται στο τέλος θα είναι ένας συνδυασμός ε, για τη διασύνδεση της Ευρώπης ε, με τα κονδύλια των διαθωτικών, κονδυλί, των ταμείων συνδέοντας αυτά με τα της ιδιωτικής δημόσιας σύμπραξης για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της ψηφιακής ατζέντα. Γιατί είναι μια καλή επένδυση. Καλό παράδειγμα. Με βάση μελέτες ε, που έγιναν για τη Γερμανία και θα έλεγα εκπροσωπώντας ε, τη Γερμανία, αυτό ισχύει και για άλλες ευρωπαϊκές αγορές και χώρες, βλέπετε ότι οι επενδύσεις ενώ είναι υψηλές με 35 δις ευρώ για αυτόν τον τομέα και βλέπετε ότι εδώ έχουμε και πρόσθετο σκέλος επενδύσεων που απαιτείται. Χρειάζεται εδώ να είμαστε ορθολογικοί, διότι θα χρειαζόντουσαν πολλαπλάσια αυτών των κονδυλίων. Βλέπετε ότι είναι καλές επενδύσεις αυτές. Γιατί, διότι με αυτές τις επενδύσεις μπορούμε να έχουμε σημαντική αύξηση στο ΑΕΠ και στις συνολικές επιπτώσεις για την αγορά είναι σημαντικότερη απήχηση σε σχέση με τις άμεσες επενδύσεις. Αν δει κανείς τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα σε σχέση με το ΑΕΠ με βάση αυτές τις ε, επενδύσεις που θα γίνουν, αυτό σημαίνει ότι οι ε, φόροι θα ε, καλύπτουν, θα αντισταθμίζουν τα ποσά αυτά τα οποία θα επενδυθούν βλέπουμε τις ε, εξωτερικές ε, ε, επιπτώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει μια σύγκληση των επενδύσεων αυτών ώστε να μπορέσουμε να έχουμε άμεσες επιστροφές από τις επενδύσεις. Επιστροφές από τις επενδύσεις. Οι εξωτερικές επιπτώσεις θα είναι πολύ ψηλότερες μοχλευτικά και αυτό δείχνει ότι η δαπάνη για τις δημόσιες επενδύσεις είναι κάτι το οποίο αξίζει πραγματικά να γίνει. Τούτων λεχθέντων εδώ θέλουμε να καταδείξουμε στη συνέχεια ότι βλέποντας το δίκτυο τηλεπικοινωνιών και επικοινωνιών είναι σημαντικό τεχνολογικά πρέπει να είναι αμερόληπτο και ουδέτερο. Θα πρέπει να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πανευρωπαϊκά. Θα έχουμε λοιπόν ε, από, ε, με τις, ε, την χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων και με κοινού κινδύνου δράσεις και επενδύσεις ιδιωτικού τομέα και κρατικού τομέα, ιδιωτικής και κρατικής σύμπραξης με τους Δήμους, τις κοινότητες ε, και στο περιφερειακό επίπεδο να υπάρξουν τέτοιου είδους ε, κοινέ ε, πρωτοβουλίες και στις υποδομές και για την δυνατότητα εκμετάλλευσης ευρύτα του φάσματος δυνατοτήτων. Βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Joint ventures με τις τοπικές κοινότητες. Θέμα ποιος θα διασφαλίζει τα κονδύλια αυτών των επενδύσεων με μεγάλες επιχειρήσεις παρόχους που ήδη επιβαρύνονται από σημαντικά χρέη που επομίζονται, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε περιόδους κρίσης ε, για να μην υπάρξει υποβάθμιση. Οι κίνδυνοι πρέπει να ε, καλύπτονται με την χρηματοδότηση αυτών των δημόσιων ιδιωτικών συμπράξεων και των πιστώσεων που θα διασφαλίζονται, μειώνοντας την έκθεση στους κινδύνους. Όλα αυτά μπορούν να συνεισφέρουν στο να μην υπάρξει διακύβευση της ε, αξιοπιστίας και της ε, φερεγγιότητάς μας όσον αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση που δεν πρέπει να διακυβευτεί. Πρέπει όλες οι δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν για την ε, διασύνδεση της Ευρώπης Connecting Europe ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Και τέλος εξίσου σημαντικό να υπάρχει ένα κερδοφόρο σκέλος το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι αποκλειστικά με πιστώσεις, θα χρειάζονται επιχορηγήσεις ε, των κρατών και του δημοσίου για να υπάρχει η πρόθεση αυτών των επενδύσεων. Χρειάζεται μια ένα, ένα ισορροπημένο, ισόρροπο μείγμα αυτών των δράσεων για την Connecting Europe Facility. Τούτων λεχθέντων όπως ήδη ε, τόνισα είμαστε πολύ ανοιχτοί για αυτήν την ε, δραστηριότητα και για τις προτάσεις που θα υποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι το Connecting Europe Facility πρέπει να συμπληρώνει παραπληρωματικά ή συμπληρωματικά αυτές τις δρόσεις και όχι να τις υποκαθιστά. Πρέπει ε, η προσοχή να δίνεται και σε μη κερδοφόρες περιφέρειες και περιοχές και να δούμε και το θέμα τη κάλυψης Τη της κερδοφορίας. Δεν είμαστε υπέρ ενός άκαμπτου, δίσκαμπτου σχεδίου ε, όσον αφορά τα μερίσματα και τις ε, επιστροφές ε, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν διάφορες περιοχές. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα των ε, περιοχών αυτών σε ένα συνδυασμό και να είμαστε ελαστικοί και ευέλικτοι. Πώς θα συνδυάσουμε τις δράσεις μας και με τις δράσεις κονδυλίων διαθροτικών ταμείων. Να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται από κοινού, συνδεδεμένα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όσον αφορά τα ειδικότερα προγράμματα, θα θέλαμε να υπάρχει και η ιδιωτικοποίηση σε συγκεκριμένο βαθμό της ε, δράσης των ταμείων και των κονδυλίων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη ε, ενίσχυσης. Θα είμαστε υπέρ του να τεθούν προτεραιότητες σε τέτοια σχέδια και προγράμματα που θα δίνουν τη δυνατότητα της χρήσης ε, συνέργειας και συνεργειών όσον αφορά τις ήδη υπάρχουσες υποδομές. Και αυτά όλα πρέπει να αντανακλώνται και στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και προτάσεων. Θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες δυνατότητες της διασύνδεσης ε, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της ε, ανάπτυξης ε, και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αύξησης του ΑΕΠ, τόνωσης του ΑΕΠ, αύξηση όσον αφορά την οικονομική δράση προς όφελος όλων των πολιτών <clears throat> με τις εφαρμογές που θα δίνουν προτεραιότητες και θα θέτουν προτεραιότητα στα σχέδια έναντι άλλων προγραμμάτων και σχεδίων υπό το πρακτικό πνεύμα εφαρμογής πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και νομική ασφάλεια και βεβαιότητα μέσω απλών κανονισμών και διατάξεων μη γραφειοκρατικού χαρακτήρα για την διαμόρφωση των χρηματοδοτικών μέσων, χρηματοοικονομικών μέσων, ιδιαίτερα ιδιωτικής και ε, δημόσιας σύμπραξης ε, για να υπάρχει η ενδεδειγμένη υποστήριξη που θα διασφαλίζεται και ε, πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για τέτοιου είδους πρόσβαση στην αγορά για το μέλλον. Ε, ε, είναι πρόσδεκτες ε, οι προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα καθορίζουν σε λεπτομέρειε με κανονισμού και διατάξεις όλες αυτές τις πτυχέ. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω εξειδίκευση των προτάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εξοικονομήσατε ένα λεπτό. Έχω μεγάλο αριθμό μιλητών και 11 λεπτά. Εισηγητέ θέλετε να πείτε τίποτα. Α, ένα λεπτό όμως ο καθένας. Τελεία. Και θα κόβω τα μικρόφωνα. Ο κύριος Ρικές. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα καταλάβανε όλοι ότι το θέμα είναι πώς ένα ιδεχθές κομμάτι κρέας θα γίνει ελκυστικό ψητό με μπόλικο σκόρδο. Υπάρχουν κριτήρια πολιτικής, ευρωπαϊκής ε, προοπτικής η προστιθέμενη αξία που είπατε και υπάρχουν καθαρά χρηματοδοτικά κριτήρια που είναι η σταθερότητα κτλ. τα κτλ. Επομένως η Κομισιόν και η ΕΤΕ θεωρούν ότι χρειάζεται να εγκαθιδρυθεί μία μεικτή δομή, μεικτή δηλαδή και αρκετά σταθερή, που να μπορεί να συνδυάσει τα χρηματοδοτικά κριτήρια, τα δημοσιονομικά κριτήρια με τα πολιτικά και δημόσια κριτήρια. Ευχαριστούμε Δομήνικε. Η κυρία Βαλιάν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Έχετε ήδη τον κατάλογο των σχεδίων και περιμένετε απλώς να το συζητήσει το Κοινοβούλιο ή όχι. Ακόμα καλύτερα. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Για τον κύριο Μέρφυ. Ο κύριος ε, Μπάιερ μίλησε για ευκαιρίες πριν από την κρίση και για το 2007. Μετά την κρίση όμως τι γίνεται, ποιες είναι οι ικανότητες, οι δυνατότητες αγοράς ε, για τις συντάξεις, για τις ασφάλειες κλπ. Για να είναι δηλαδή ενεργές σήμερα. Στον κύριο Πακέ, η κεντρική διαχείριση, τι, ε, τι, καλό και τι κινδύνους ε, θα, θα, θα είχε για την χρηματοδότηση και τι θα ήταν, ποιος θα διαχειριζόταν το εκτελεστικό κέντρο για τα δίκτυα. Και για τον κύριο Ντάουλ μίλησε για την αύξηση του ΕΠ. Θα μπορούσατε εσείς από τις ε, τηλεπικοινωνίες ε, να θέσετε συνέργεια για τις μεταφορές, γιατί όλα αυτά γίνονται μέσα σε πολύ κλειστά ε, πλαίσια. Ντεμπάκερ, ευχαριστώ. Τρει ερωτήσει. Η ερώτηση ήδη τοποθετήθηκε για το crowding out effect. Η ίδια ερώτηση θέλω να θέσω. Υπάρχει ένα τέτοιο κίνδυνο. Πώ μπορεί να διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα υπάρχει τέτοιο φαινόμενο. Μετά, για τι επικρίσει για του οίκου πιστοληπτική αξιολόγηση, πρέπει να περιμένουμε να δούμε, είπανε, πώ θα διαμορφωθούν αυτά τα προγράμματα για να κρυθούν οι πιστοληπτικέ αξιολογήσει όσον αφορά τα ομόλογα. Έχετε κάποιε απόψει από αυτού. Τελευταία ερώτηση όσον αφορά, κύριο Πακέ. Ξέρω ότι σε σχέση με τη διαμόρφωση απόψεων στον τομέα των μεταφορών. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι υπό την τεχνολογική προοπτική θα υπάρχει ουδετερότητα και αμεροληψία και θα υπάρχει η εγγύηση, ε, υπάρχει πολλή έμφαση στα σιδηροδρομικά δίκτυα ή στα οδικά δίκτυα. Τι μπορεί να γίνει σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κράμερ, ένα λεπτό τώρα παρακαλώ. Όχι εσείς, η κυρία Λίχτενμπέργκερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και πάλι για άλλη μια φορά τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ρωτήσω ποιο είναι το επίκαιρο τμήμα μεταξύ σιδηροδρόμων και οδικών δικτύων και inland waterways των εσωτερικών ε, ποτάμεων ε, αρτηριών ε, διασυνδέσεων. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Φαίνεται το τομέα των οδικών μεταφορών είναι πολύ υψηλότερο. Δεύτερον, το υψηλότερο ποσοστό των οδικών, του οδικού τμήματο οφείλεται στην ταχύτερη υλοποίηση και ε, ε, δυνατότητα ολοκλήρωσης και από την δομή τελών και ε, εσόδων που μπορούν να εισπράττονται. Είναι εδώ τουλάχιστον και το θέμα της συντήρησης και διατήρησης δικτύου που συνεισφέρει. Δεύτερον, πώς μπορούν και τα κριτήρια του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά κριτήρια να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βουίτς, παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση προς εμάς, κύριε. Ποιο τμήμα θα είναι η κάλυψη κινδύνων μέσω των ε, ομολόγων έργου από την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων και για ποιο χρονικό, ε, ποια χρονική διάρκεια και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η κερδοφορία όταν δεν είναι γνωστά αυτά τα στοιχεία και όταν υπάρχει και κίνδυνος που διαγράφεται εδώ για μια τριαντακοντή Λοιπόν, ε, περίοδο μπορεί να υπάρξει κάποια ένδειξη και τι γίνεται σε σχέση με την επαναχρηματοδότηση των οδικών τέτοιων σχεδίων χρειάζονται επιπρόσθετα για την διασφάλιση, για την κατοχήρωση των ιδιωτικών ε, κερδών ε, έσοδα τα οποία θα προβλέπονται από τα τέλη που θα καταβάλουν αυτά τα ε, ιδιωτικά οχήματα. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Πακέ. Μας είπατε ότι οι επενδυτές και επενδύτριες χρειάζονται καλύτερα προγράμματα. Μέχρι τώρα είχα καταλάβει ότι τα πολυάριθμα προγράμματα που επεξεργαζόμαστε εδώ και 15 χρόνια ήταν όλα καλά και ότι απλώς η χρηματοδότηση έλειπε. Πώς κρίνετε λοιπόν τα προγράμματα αυτά, τα θεωρείτε μέτρια, κακά, με εντυπωσίασε αυτή, αυτό που είπατε. Τι αναμένεται κατάλογος καλών προγραμμάτων και τώρα για τον κύριο Μέρφη και την ΕΤΕ. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως βουλευτές για να αυξήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης δανειοδοτήσεων από την ΕΤΕ που είναι περιορισμένες. Τα 50 δισεκατομμύρια προτείνει Κομισιόν Είπαμε ότι ίσως να είναι και ανεπαρκή. Οι δυνατότητες δανειοδότησης της ΕΤΕ μπορούν να επεκταθούν και πώς. Κυρία Μάισνερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι τα πιλωτικά προγράμματα. Γνωρίζουμε επίσης ε, ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις πολλές φορές σε τέτοια ε, προγράμματα. Γι' αυτό, τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρέπει να εγκριθούν οι όροι και προϋποθέσεις ε, πλαίσια για αυτές τις δράσεις, αλλά παράλληλα πρέπει να προετοιμαστούν με την Ευρωπαϊκή, Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά. Ποια προγράμματα θα είναι αυτά για να πιστούν τα κράτη-μέλη. Βράχει πρόθεσμα να πιστούν ότι τέτοιου είδους πιλωτικά προγράμματα μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Σε ποιο βαθμό έχετε προχωρήσει. Υπάρχουν πιθανοί επενδυτές με τους οποίους να είσαστε σε επαφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κράμερ ένα λεπτό τώρα. Λοιπόν, το ότι αυτά τα μεγάλα προγράμματα για τις τράπεζες, για τις οικοδομικές εταιρείες είναι θελκτικά, είναι θελκτικά γιατί άλλοι τα πληρώνουν. Εντάξει, αλλά όριο. Πού βρίσκεται, ερώτηση, πού βρίσκεται εδώ το όριο για την χρηματοδότηση σε σχέση με, τα, με αυτά που γίνονται στην ε, Γερμανία και αυτά που γίνονται στην Γαλλία. Χάλε, ε, Νιρεμβέργη με πολλές ε, σύραγγες ε, που συνεπάγεται πολλές δυσκολίες ενώ Λάιψιχη Χιγένα θα ήταν μια καλύτερη διασύνδεση το ίδιο Βιέννη Γκράτς προς την Αδριατική θάλασσα που είναι πάρα πολύ δαπανηρό εγχείρημα και την, έχουμε και την Πανωνική Κοιλάδα που θα ήταν μια εναλλακτική δυνατότητα. Πού βρίσκονται τα όρια για όλα αυτά. Αναφέρθηκαν τα σταθερά κόμματα εδώ έχουμε πυρηνικό αντιδραστήρα για την ε, Φινλανδία. Τι γίνεται με τους κινδύνους από πλευράς του δημοσίου. Έχουμε σύραγγες ε, ε, έργα τέτοια τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Τι γίνεται με αυτά. Ευχαριστώ. Κάντσαν παρακαλώ ένα λεπτό. Σύντομα. Κύριε Πακέ, άμα μείνουμε εμείς μέσα στο ΣΥΕΦ και το 80% το μοιράζουμε ως γκρέντ... Είναι άχρηστο να μιλάμε για νέους μηχανισμούς, πολλαπλωσιαστικούς παράγοντες ή οτιδήποτε άλλο. Άμα ξεπεράσουμε όμως το όριο της EF, έχουμε και άλλες δυνατότητες ε, για να, κάνουμε, να αναπτύξουμε όλα τα σκεπτικά που αναφέραμε σήμερα το πρωί, γιατί αλλιώς εδώ κοροδιευόμαστε. Θα θα ήμουν ευγνώμων στους διερμηνείς άμα μας δίνανε 5-6 λεπτά παραπάνω. Δύο λεπτά τώρα οι ομιλητές. Αν δεν καταφέρετε να απαντήσετε σε δύο λεπτά μπορείτε να στείλετε email ή και πιστολές ακόμη αν θέλετε. Ευχαριστώ για τι εξαιρετικέ ερωτήσει. Το δυνατόν συντομότερα χρηματοοικονομικά κριτήρια για τι δράσει τη τράπεζα που αξιολογούνται οικονομικά και που περιβαλλοντικά εγκρίνονται, δηλαδή με άλλα λόγια ανταποκρίνονται σε κριτήρια. Χρηματοδοτεί προγράμματα η τράπεζα που ευθυγραμμίζονται με τι προτεραιότητε των εθνικών αρχών και των ευρωπαϊκών αρχών ω προτεραιότητε. Τώρα, crowding out effect πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντική χρηματοοικονομική ανάγκη επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο, αλλά υπάρχει και ρόλος και για άλλους. Βλέπουμε ένα καταλητικό μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει η αύξηση μεριδίων άλλων που θα εμπλέκονται. Πιλωτικά προγράμματα και αξιολογήσεις πιστοληπτικές. Ναι, οι ε, οίκοι αξιολόγησης υποβάλλουν ε, άποψη και σύσταση για τέτοιου είδους προγράμματα. Εμείς ε, χρησιμοποιούμε τέτοιες αξιολογήσεις και θα υπάρχει η συνέχιση αυτών των δραστηριοτήτων. Μετά, πρωτοβουλία ομολόγων έργου σε σχέση με την δομή και την ε, ανάπτυξη έργου. Για το 20% για παράδειγμα ε, κάλυψης ε, κινδύνου που λαμβάνεται υπόψη για, ως κατευθυντήρια γραμμή για προγράμματα τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη. Διατήρηση, συντήρηση και περιβαλλοντικά κριτήρια διατήρηση συντήρηση ε, όσον αφορά την πτυχή αυτή πρέπει να έχουμε ένα, μια σαφή ένδειξη δέσμευσης όσον αφορά την συντήρηση, διατήρηση. Δεν έχει νόημα να επενδύονται χρήματα σε προγράμματα τα οποία μπορούν να καταρρεύσουν ή μετά διαβρώνονται επειδή δεν υπάρχει συντήρηση, ε, διατήρηση. Όσον αφορά την πρωτοβουλία ομολόγων έργου, ε, περνά μέσα από την διαδικασία ε, αξιολόγηση έγκρισης. Ο μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί για την, απόσβεση, για την κάλυψη κινδύνων μέσω του μέσου που περιγράφει και πιο πριν. Και με αυτή τη βάση μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Τι μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμα τι μπορεί να ε, γίνει για να διευρυνθεί αυτή η δραστηριότητα. Υπάρχει ευρύτερη συζήτηση για τα κεφάλαια κινδύνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνδέοντας τα, τα χρηματοοικονομικά μέσα σημαντικότερο μέσο για την χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. 10% αυτό είναι μεγάλη εξοικονόμηση όσον αφορά τις τράπεζες. Εσείς παρακαλώ ε, μπορείτε να παρέμβετε. Ναι, χρειαζόμαστε καλύτερα ενωσιακά προγράμματα και προγράμματα με μεγαλύτερη ευθυγράμμιση για στις ανάγκες των μεταφορών και καλύτερα δομημένα για να ελκύουν και η δημόσια και η ιδιωτική χρηματοδότηση. Επομένως, η υπηρεσία που περιγράφω θα βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία των προγραμμάτων και στην καλύτερο μηχανισμό επιλογής τους. Φυσικά δεν είναι παρά ένα εργαλείο. Η Κομισιόν θα παραμείνει βασικός παράγοντας και άλλες υπηρεσίες και όργανα θα παίξουν ρόλο και σε συνεργασία με την ΕΤΕ και άλλες υπηρεσίες και όργανα θα υπάρξει επιτέλους ένας μηχανισμός καλύτερης προετοιμασίας και όπου θα μπορούσαμε να λύσουμε το τετραγωνισμό του κύκλου που ανέφερε ο Δομήνικος Ρικέ. Δηλαδή και καλύτερη προετοιμασία των πιο ενωσιακών προγραμμάτων και τέτοιου είδους προετοιμασία με τον συνδυασμό δημοσίου και ιδιωτικού χρήματος ώστε να μπορεί η ΕΤΕ να συμπληρώσει τις ελλείψεις αν διαπιστωθούν. Έχουμε κατάλογο προγραμμάτων, πολύ λεπτομεριακό. Στην προσθήκη 1 και στο ICT και για την ενέργεια. Αλλά εκεί πρέπει να συμπληρωθούν οι κατάλογοι δεν μπορώ τώρα να σας τα παριθμίσω όλα, αλλά φυσικά υπάρχουν, θα τα μάθετε και είναι σε συνεννόηση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Βερικά από αυτά απαιτούν περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση από ό,τι άλλα. Δεν έχουν όλα την ίδια μίξη. Ευχαριστούμε. Ντόλ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ρώτησαν Ποιο είναι ο συνδυασμό ακριβώ των ενεργειακών προβλημάτων με τι μεταφορέ. Οι συνδυασμοί που θα μπορούσαν να γίνουν οι συνέργειες είναι ότι περίπου 8% αφορά δημόσια έργα, ένα τρίτο είναι η αξιολόγηση κτηρίων και λειτουργικού κόστους και στη Γερμανία ιδιαίτερα έχουμε μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία με τοπικές αρχές για τα δημόσια έργα. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο το συντονισμό και τη συνεννόηση μειώνονται το κόστος πράγμα που σημαίνει αύξηση της αποδοτικότητας των προγραμμάτων και φυσικά μεγάλη επέκταση του εύρους εφαρμογής αυτών των σχεδίων. Είναι πολύ σημαντική διάσταση λοιπόν. Καλύτερος μηχανισμός συντονισμού, η καλύτερη χρήση της ενέργειας για τα κτίρια και, και την κατασκευή μάλλον των δικτύων, καθώς και καλύτερη χρησιμοποίηση των υπαρχουσών υποδομών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από πολλαπλούς τομείς Βέβαια ο καθένας τον τομέα του γνωρίζει και θα μπορούσαν να γίνουν και συνδυασμοί και έτσι να χαμηλώσει ακόμα περισσότερο το κόστος και η ανάγκη δημόσιας χρηματοδότησης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τα μέλη και τους ομιλητές και ομιλήτριες και του δεύτερου γύρου που με βοήθησαν να σεβαστώ το χρονοδιάγραμμα. Και τώρα ξαναδίνω το λόγο στον προηγούμενο, στην προηγούμενη πρόεδρο. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες και τους διερμηνείς. Η Ήτρε θα ξανασυνεδριάσει στις 3. Ευχαριστώ και τους εισηγητές.